Colleagues, please be seated. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Να ξεκινήσουμε απευθείας. Κοινή δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας για την εφαρμογή της ε, ρήτρα αλληλεγγύης. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μωράες, πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για να μας κάνει ορισμένα εισαγωγικά σχόλια. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση των μελών ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Καθυστερήσαμε με την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ζητώ και πάλι συγγνώμη. Συνάδελφοι, από πλευρά Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και να ευχαριστήσουμε και την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και την Πρόεδρο για την πρόσκληση. Σας καλωσορίζω όλους σε αυτήν την κοινή κρόαση για την εφαρμογή της ρήτρα αλληλεγγύης που συνδιοργανώνεται από τις δύο επιτροπές. Είναι ικανοποιητικό ότι αυξάνεται ο αριθμό των κοινών ακροάσεων με άλλε επιτροπέ και σήμερα το πρωί είχαμε κοινή δημόσια ακρόαση με την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου για τις ροές δεδομένων και αυτό αυξάνει τις δυνατότητες ε, για την Επιτροπή μας να κατανοήσει τι συμβαίνει και με το έργο άλλων Επιτροπών. Αυτό συμβαίνει και εδώ σήμερα. Τα θέματα που εξετάζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο είναι ε, οριζόντια και διατομεακά. Το σημερινό ζήτημα είναι πολύ γνωστό και σημαντικό. Η ρήτρα της αλληλεγγύης και εγώ το έχω δει εδώ και πολλά χρόνια γιατί είμαι στο κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια. Είναι θέμα ιδιαίτερα προσφυλέ ε, και σε εμά και στου ε, πολίτε μα και στι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Η ρήτρα αλληλεγγύη που εγγράφεται στο άρθρο 22 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να υπάρχει κοινή ανταπόκριση των κρατών μελών εν ώψη ε, φυσικών καταστροφών, ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών επιθέσεων κ.ο.κ. Και εφόσον όλα αυτά συμβαίνουν ε, με αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ξέρουμε ότι ε, η σύλληψη αυτού του άρθρου έχει μακρά ιστορία και ήταν επαναστατική η αρχική ιδέα, ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη είναι πρωταρχικά υπεύθυνα για τη διαχείριση κρίσεων εντός ε, της επικράτειάς τους, ιδίω μεγάλη κλίμακα, είτε φυσικέ είτε ανθρωπογενεί καταστροφέ, που είναι διασυνοριακέ πολύ συχνά, διατομιακέ και ξεπερνούν τι επιμέρου δυνατότητε ενό κράτου μέλου. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, απαιτείται κάποιο είδου ρήτρα αλληλεγγύη. Και αυτό αποτέλεσε την απαρχή αυτή τη ρήτρα. Πέρυσι, στι 24 Ιουνίου 2014, κατόπιν μακροσκελού συζήτηση και διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο υιοθέτησε ε, απόφαση για την εφαρμογή της ε, ρήτρας αλληλεγγύης της Ένωσης η σημερινή ακρόαση θα εξετάσει την βραχυπρόθεσμη πρακτική εφαρμογή του άρθρου αυτού, δηλαδή τη θέσπιση και αξιοποίηση των διευθετήσεων που υιοθετήθηκαν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2014 σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της ε, ρήτρας αλληλεγγύης, της ανταπόκρισης σε ενωσιακό επίπεδο και της αξιολογήσης απειλών σε ενωσιακό επίπεδο. Προς το παρόν, ε, περισσότερο επί χάρτου υφίσταται αυτή η ρήτρα, από όσο γνωρίζω εγώ, κανένα κράτο μέλο δεν έχει ζητήσει και δεν έχει επικαλεστεί την ρήτρα τη αλληλεγγύη, όμω με ενδιαφέρον θα ακούσω και του ομιλητέ μα. Θα ήθελα εδώ να ακούσουμε πώς εκείνοι ε, βλέπουν τη σύνδεση της ρήτρα αλληλεγγύη και άλλων μηχανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Ανταπόκρισης κρίση και αν υπάρχουν άλλα συγκεκριμένα κριτήρια για την επίκληση της αρχής της ρήτρας αλληλεγγύης. Πολλά ακόμα ζητήματα θέλω να θίξω, αλλά εφόσον καθυστέρησα δεν θέλω να μακρηγορήσω. Έχουμε πολύ διακεκριμένους ε, ομιλητές ε, σήμερα μαζί μας. Είναι και απόγευμα, είμαστε όλοι κουρασμένοι, επομένως ε, θα μείνω εδώ και να δώσω το λόγο στη συμπρόεδρο Άννα, πρόεδρο της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας, για τα δικά της εισαγωγικά σχόλια και βεβαίως να παρουσιάσει τους ομιλητές μας. you very much Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Δεν θα ήθελα να σπαταλήσω πολύ χρόνο. Απλά θα συμφωνήσω με τα λόγια του συναδέλφου ότι η ρήτρα αλληλεγγύης είναι ελάχιστα γνωστή μετά από ένα χρόνο και την απόφαση του Συμβουλίου υπάρχει κάποια παρανόηση της ε, ρήτρα αυτής. Ε, θα ήθελα λοιπόν οι προσκεκλημένοι μας ε, να συζητήσουν, να μας μιλήσουν για αυτό το ζήτημα. και να μας πούν ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις ε, δύο ρήτρε. και τώρα να σας παρουσιάσω τους ε, διακεκριμένους προσκεκλημένους πρώτον πρόσωπος της Προεδρίας είναι ο κύριος Ούντις Μίκουτς πρόεδρος των φίλων της Προεδρίας και ασχολείται με θέματα που αφορούν την ανταπαντήσεις στις πολιτικές κρίσεις. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το ζήτημα αυτό που είναι ελάχιστα γνωστό Δεύτερον, ε, δεύτερος εξαριστερός μου, ο κύριος Χάνς Ντάς από την ε, Κομισιόν, ε, συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Και έχουμε και άλλους δύο εμπειρογνώμονες, τον κύριο Νίλς Μπρακέ, που εκπροσωπεί το Κέντρο Πληροφοριών και ο κύριος Ρόντερικ Πάρκς από το Σουηδικό Ινστιτούτο Διεθνών ε, ε Υποθέσεων και δώσω τον λόγο πρώτα τον κύριο Μίκουτς και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι. Παρακαλώ κύριε Μίκουτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό από μεσήμερο. αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να απευθύνομαι προς εσάς επί ενός τόσο σημαντικού ζητήματος. Εάν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει διερμηνία, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά και να εκμεταλλευτώ τις γνώσεις μου για να μπορέσετε να με καταλάβετε πιο άμεσα. Συνεχίζω λοιπόν ε, στα αγγλικά. Δεν θα ήθελα να σας ζαλίσω με πολλά λόγια σχετικά με το περιεχόμενο του ΑΡΘΟΥ 22 για τη ρήτρα αλληλεγγύης και για την απόφαση του Συμβουλίου περιφαρμογής αυτής θα ήθελα να εστιάσω την παρέμβασή μου στο πνεύμα που βρίσκεται πίσω από τις ε, αποφάσεις που έχει λάβει το Συμβούλιο και θα ήθελα να ανοίξω το δρόμο για περισσότερες ανταλλαγές ε, απόψεων επί του ζητήματος. Δεδομένου το ότι οι καταστάσεις που καλύπτει η Ρήτρα απαιτούν ε, από όλους τους θεσμούς να συνεργαστούν. Φυσικά πρόκειται για την αλληλεγγύη, αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και αλληλεγγύη που εκφράζεται μέσω των θεσμών της Ένωσης σε περίπτωση που ένα από τα κράτη-μέλη γίνει ε, αντικείμενο κάποιες τρομοκρατικής επίθεσης ή υποστεί κάποια σημαντική καταστροφή. Αυτό είναι κάτι που αφορά την ικανότητα των κρατών μελών για ανταπόκριση σε παρόμοιες καταστάσεις. Η ρήτρα αλληλεγγύης δεν αντικαθιστά κάποιο άλλο ενωσιακό εργαλείο αλλά προσπαθεί να δυναμώσει τα ισχύοντα εργαλεία και μέσα. Να σας πω τώρα με μερικές προτάσεις πώς καταλήξαμε στην προσέγγιση. Το άρθρο 222 δεν είναι από τα πιο σαφή άρθρα της συνθήκης και μια σειρά από ζητήματα έπρεπε να διευκρινιστούν περαιτέρω και να αναλυθούν από νομική σκοπιά. Φυσικά τα εγκάρσια ζητήματα αυτού που αφορά, αφορούν σε αυτό το άρθρο απαιτούν μια καινοτόμο και κλαδική προσέγγιση, πολυκλαδική προσέγγιση. Γι' αυτό και η ομάδα φίλων του Προεδρίας το οποίες εγώ προεδρεύει, προσπαθεί να διασφαλίσει την κατάλληλη διαχείριση αυτών των κοινών προτάσεων, πώς να προωθηθούν. Μετά από μια σειρά ε, συναντήσεων, το ζήτημα διευθετήθηκε και το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση με ομοφωνία. Να τράξω την ευκαιρία λοιπόν για να ευχαριστήσω και το Ευρωκοινοβούλιο για την σύμβολή του για την έκθεση του 2012 αναφορικά με τη ρήτρα αμοιβαίας ε, αλληλεγγύης. Επανδημένα το, και το Συμβούλιο μόνο κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν πως η ρήτρα αλληλεγγύης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές έκτακτες περιστάσεις όταν όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέσα έχουν καταδειχθεί ανεπαρκή. και μια τέτοια ρήτρα απαιτεί έναν ύψιστο βαθμό πολιτικής συνεργασίας. Το Συμβούλιο όμως ε, τήρησε τις ε, αρμοδιότητες των ε, ενωσιακών υπηρεσιών. Στόχος ήταν να υπάρξει μια συνεκτική, ένα συνεκτικές και ολοκληρωμένο σύστημα. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, επιτευχθεί αυτό πρώτα απ' όλα. Θέλαμε το Συμβούλιο Εξωτερική Επιτροπή και, και η Κομισιόν συγγνώμη, θα έπρεπε να έχουν την αυτή προσέγγιση. Τώρα, αυτό μεταφράζεται σε μια προσέγγιση που αφορά μια έγκαιρη συμμετοχή του Συνοβουλίου και να μην αναθέτει καμία ευθύνη ε, προς την Κομισιόν και την είπα εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Θα ήθελα να τονίζω πως το Συμβούλιο θα εστιάσει σε μια πολιτική ανταπόκριση, πολιτική απόκριση. Σε επιχειρησιακό επίπεδο θα υπάρξει ένα συντονισμός από το αρμόδιο κέντρο και ο συνάδελφός μου Χάνιστο θα σας μιλήσει σίγουρα περισσότερα αργότερα. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο, αλλά σημαντικό, Αυτός είναι ένας μηχανισμός κρίσης σχετικά νέος που επιτρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και να ε, δώσουμε μία απάντηση άμεσα και τάχιστα στην κατάσταση της κρίσης. Αξιότιμα μέλη. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί θεωρητικό, αλλά να σας ε, μιλήσω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη αν η ρήτρα αλληλεγγύης επικληθεί. Ας σκεφτούμε μια περίπτωση όπου εμπλέγεται ένα κράτος μέλος που ε, θα μπορούσε να αφορά την έκρηξη ενός ηφαιστείου όπως συνέβη στην Ισλανδία ή πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις. Έτσι το κλειέν κράτος μέλος είναι ο πρώτος ε, ε, αποκριτής. Η ρήτρα αλληλεγγύης προοδευτικά έχει ήδη εφαρμοστεί μέσω της κινητοποίησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και ούτω καθεξής, αλλά εάν τα διαθέσιμα μέσα στη χώρα είναι ανεπαρκή, ό,τι κατά κυβερνήσεων ο Πρωθυπουργό ή ο Πρόεδρο τη χώρα μπορεί να ζητήσει, να προβεί σε επίκληση τη ρήτρα αλληλεγγύη. Για να διασφαλίσουμε μια γρήγορη κινητοποίηση των ενωσιακών πόρων θα πρέπει να υποβληθεί γραπτός το αίτημα και στον πρόεδρο της Κομισιόν μέσω του κέντρου εκτακτής ανάγκης και θα υπάρξουν άμεσες συνέπειες Ας δούμε λοιπόν ποια διαδικασία που Πρώτον, εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί, BCR ε, ή ε, ο μηχανισμός κρίσης θα ενεργοποιηθεί άμεσα και αυτό θα οδηγήσει σε αποστολή ε, ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα κράτη-μέλη ή στην Κομισιόν και στον Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης. Και εδώ προβλέπεται μια κάποια πλατφόρμα την οποία ε, διαχειρίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου ως Προεδρία. Θα έρθει σε επαφή με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου προκειμένου να ενημερωθεί για την επίκληση. Ίσως ε, αργότερα ο μόνιμος εκπρόσωπος ε, να συγκαλέσει μια στρογγυλή τράπεζα για να δει κατά πόσο το Συμβούλιο μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει τον συντονισμό. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτική Δράση εμπειρογνώμονοι και άμεσα ενδιαφερόμενοι εμπλέκονται στην υπόθεση. Και φυσικά ο συντονιστής θέματα τρομοκρατίας πρόκειται για θέμα, ζήτημα τρομοκρατίας. Στόχος είναι να είμαστε σε καλύτερη θέση και να έχουμε καλύτερη ενημέρωση για να αποφασίσουμε για τις ε, εργασίες που να εξαχθούν περαιτέρω. Και μπορεί να συγκληθεί εντός ορών μια συνεδρίαση και αυτό θα εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα των ε, Υπουργών αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν θα γίνει τίποτα ε, είπατε εκπρόσωπος ε, Ιστορικής Πολιτικής Ένωσης θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις οι υπηρεσίες προσπαθήσουν να προετοιμάσουν την κοινή ολοκληρωμένη έκθεση προκειμένου να ενημερώσουν και να δώσουν μια κατάλληλη εικόνα τη κατάστασης. Παρόμοιες εκθέσεις θα είναι διαθέσιμες την επόμενη μέρα. Ευθύς αμέσως ε, συγκαλεί ο Πρόεδρος ε, μια συνεδρίαση για να εξετάσουν την κατάσταση και ούτω καθεξής. Ε, τέτοια παρόμοιες συζητήσεις χρησιμεύουν για δημιουργία καλύτερων συνεργειών και καλύτερο συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων. Στο τέλος ε, το Συμβούλιο αφού λάβει αποφάσεις ε, η πλατφόρμα του κέντρου χρησιμοποιείται ως ε, γραμματεία για την πρόθεση πληροφοριών και αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί. Αξιότιμα μέλη εργαζόμαστε με, στο Συμβούλιο με την υποστήριξη της Κομισιόν και της ΥΠΑΤΗ ε, ε, της ύπαντης εκπροσώπου. Προσπάθησα να σας εξηγήσω πώς ε, θα έχει η κατάσταση. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για αλληλεγγύη. Όταν υπάρχει μια κατάσταση κρίσης, σε παρόμοιες καταστάσεις δεν μπορούμε να μην έχουμε υπόψη τις απαιτήσεις των πολιτών. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι χέρι-χέρι ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του καθενός. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο όντω είναι κρίσιμο στο πλαίσιο όπου οι καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προετοιμαζόμαστε με τον, καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Είναι το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αντιμετωπίζει τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας εκτός της Ευρωπαϊκής αλλά και τα θέματα προστασίας των πολιτών στο ιστορικό και το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχειριζόμαστε λοιπόν τον ε, μηχανισμό προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ένα όργανο το οποίο, ένα εργαλείο το οποίο υφίσταται πλέον 10-15 χρόνια και έχει αποδεχτεί ιδιαίτερα επιτυχίες σε ό,τι αφορά την συντονισμό των ε, κρατών μελών σε θέματα ανταπόκριση σε τέτοιε καταστάσεις. Θα ήθελα να προσθέσω στην εικόνα που με μεγάλη λαφυρότητα μας παρουσίασε ο προηγούμενος ομιλητής την ε, άποψη και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του Κέντρου Συντονισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που ε, είναι υπό την εποπτεία της DG ECO. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η ρήτρια αντιλεγγύης και η εφαρμογή της δεν ε, ε, ισχύει εν κενό. Πολλά, διάφορα εργαλεία, πολλά και διάφορα εργαλεία υφίστανται ε, εδώ και χρόνια για την αντιμετώπιση κρίσεων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και η συνολική προσέγγιση η οποία επιλέχτηκε εξ αρχής για την ανάπτυξη της ρήτρας ε, αλληλεγγύης και των εφαρμοστικών κανόνων ήταν ότι θα βασιστούμε ακριβώς αυτά τα υφιστάμενα μέτρα και εργαλεία για να στηριχθούμε στο βαθμό του δυνατού σε αυτά που ήδη υπάρχουν και ήδη έχουν αποδεχτεί ότι λειτουργούν καλά. Η εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης έπρεπε να είχε ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού μάλλον των μέτρων αυτών. Επίσης, ε, πολλοί από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων μας είπαν λίγο πολύ ότι δεν υπήρχε επιπρόσθετος ε, προϋπολογισμός ε, και επιπρόσθετη χρηματοδότηση και θα έπρεπε να στηριχθούμε σε αυτά τα μέσα που ήδη υφίστανται. Άρα δεν υπάρχουν νέες δομές, απλά προσπαθήσαμε να συντονίσουμε τις ήδη υφιστάμενες δομές. Άρα ουσιαστικά η ρήτρα αλληλεγγύης μας δίνει ένα καινούργιο πλαίσιο, πλαίσιο για καλύτερη δουλειά, καλύτερη συνεργασία βάσει των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων, εργαλείων, μέσων, θεσμικών ρόλων και Τι είναι λοιπόν η ρήτρα αλληλεγγύης συμπερασματικά. Προφανώς δεν προορίζεται για την ε, ε, ετήσια πλημμύρα, την ετήσια πυρκαγιά στα κράτη-μέλη. Τέτοιου είδους καταστροφές, όσο δύσκολες και δραματικές και αν είναι, αντιμετωπίζονται από τον κανονικό μηχανισμό προστασία των πολιτών ή από άλλα εργαλεία τα οποία διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που συζητάμε είναι εξαιρετικέ περιπτώσει, καταστάσει που πραγματικά ξεπερνούν κατά πολύ τι κανονικέ ε, ακόμα και μετά την εξάντληση των πόρων και των μέσων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Κάποια από τα σενάρια τα οποία έχουμε επεξεργαστεί είναι Απλό για παράδειγμα, στην πόλη της Νάπολης έχουμε το Βεζούβιο, το Ηφαίστειο και η έκρηξη ε, είναι μία φορά στα 2.000 χρόνια. Αν αυτό συμβεί αύριο, όλη η πόλη της Νάπολης θα καταστραφεί και μιλάμε για εκατομμύρια άνθρωπους, ανθρώπους που θα χάσουν την κατοικία τους. Αυτό προφανώς θα υπερφορτώσει τις εθνικές ικανότητες της κάθε χώρας και ασφαλώς και θα ξεπεράσει τα εργαλεία που έχουμε ήδη σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα χρειαστούν λοιπόν επιπρόσθετα μέσα, επιπρόσθετη βοήθεια. Για παράδειγμα, τροποκρατική επίθεση, χημική επίθεση, μία, ένα τύχημα τύπου Τσέρνομπιλ με μόλυνση αλλά και μαζική α, εκένωση πολιτών. Μιλάμε για καταστάσεις στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Η αιτία Τη ε, κρίση θα μπορούσε να είναι και εκτό των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Για παράδειγμα, μια τρομοκρατική επίδοση στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντίκτυπο όμω στο εσωτερικό τη επικράτεια. Και σε κάθε περίπτωση μιλάμε για την κινητοποίηση πολλών φορέων. Διατομεακή κινητοποίηση. Γιατί τέτοιου είδου περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν φορέα, από μία αρχή μόνη τη, Πάντα προαπαιτούν οριζόντια συνεργασία, συντονισμό όλων των φορέων σε επίπεδο κράτους μέλους αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνει και κάποιες από τις τρεις χώρες, κάποιους εταίρους, διεθνείς, οργανώσεις, μη κρατικούς φορείς. Κοινωνικά μέσα μαθαμένα και, και αυτά μαθαμένα τα χρησιμοποιούμε γιατί πραγματικά δραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε τις καταστάσεις. Τι θα κάνουμε λοιπόν σε μια κατάσταση τέτοια σε ό,τι αφορά και την ρήτρα αλληλεγγύης. Θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας τα υφιστάμενα μέσα για να αξιοποιήσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία. Ε, σίγουρα ένα εξ αυτών θα είναι και ο μηχανισμός προστασίας των πολιτών, αλλά και κάποια εργαλεία των ε, συναδέλφων στη Γενική Διεύθυνση Υγείας σε ό,τι αφορά επίσης τα ε, μέσα καταπολέμησης τρομοκρατίας από τη Γενική Διεύθυνση Home και έτσι λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασικά θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα συντονιστούν η χρήση και θα είναι βέλτιστη η χρήση των μέσων αυτών. Και σε κάθε περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είναι επαρκή τα μέσα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενδεχομένω να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον θεωρούνται επαρκή τα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να προτείνει επιπρόσθετα μέτρα, να, καταβάλει, να καταθέσει δηλαδή νέε προτάσει σύμφωνα με τα θεσμικά ισχύοντα μέτρα. Αποκινούμε την είπατε εκπρόσωπο σε, κάθε, σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά τα επιπρόσθετα λοιπόν μέτρα, τι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν fast tracking για την έγκριση νέων φαρμάκων, για παράδειγμα γρήγορη τροπολογία, τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας για να γίνει απαλλαγή από τέτοιες ε, απαιτήσει. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία με την καταστροφή στη Φοκουσίμα, όταν αντιμετώπισε την καταστροφή λοιπόν αυτή, τις πρώτες έξι εβδομάδες μετά το ατύχημα, χρειάστηκε να τροποποιηθούν 150 ε, εθνικά νομοθετήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για το νομοθέτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα μας περίμενε εμά, στην Ευρώπη σε διάφορα επίπεδα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχομένως να χρειαστεί να συμμετάσχει και να αναμειχθεί σε νομοθετική διαδικασία. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να έρθουμε στο ύψο των περιστάσεων και να συνεργαστούμε. Το ERCC, το Κέντρο Ανταπόκρισης και συντονισμού σε περιπτώσεις κατεπίγουσας ανάγκης ERCC αποτελεί το βασικό κόμβο όπου θα συγκεντρωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες ή πιο πολλές εξ αυτών. Να σας πω λοιπόν δύο λόγια για αυτό το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε επισκεφθεί. Αν το έχετε επισκεφθεί, σας καλώ θερμότατα να το επισκεφτείτε. Είμαστε κέντρο ανοιχτό με ιδιαίτερη διαφάνεια. Ίσως θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε λοιπόν ε, μια κοινή επίσκεψη των δύο επιτροπών ε, με κάποια καθοδήγηση από πλευρά μα. Είναι καινούργιο το κέντρο λοιπόν αυτό. Ένα κέντρο αντιμετώπιση κρίσεων με μεγάλη διαφάνεια. Δεν είναι σημείο α, οχυρωμένο. Είναι ένα μέρος για τη συλλογή πληροφοριών ε, αποτελείται από διάφορα γραφεία σε διάφορα σημεία των Βρυξελών στα οποία μπορεί να μεταβεί κανείς για την ανταλλαγή πληροφοριών. Το ERCC λοιπόν αποτελεί το αρχηγείο συντονισμού όλης, ε, όλη του όγκου εργασίας για την προστασία πολιτών, για την ανθρωπιστική βοήθεια και ε, σταδιακά καθίσταται πλατφόρμα κρίσεων για διάφορε άλλε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει οριζοντία υποστήριξη σε πολλέ γενικέ διευθύνσει. Σε ό,τι αφορά την ε, επίκληση τη ρήτρα αλληλεγγύη, θα δρούσαμε λοιπόν ω κέντρο συντονισμού και ω σημείο εισόδου. Οποιαδήποτε αίτημα από τον πρόεδρο τη Επιτροπή θα γινόταν μέσω του ERCC, λοιπόν, στην υποθετική περίπτωση ε, κρίσης. Και θα ήμασταν λοιπόν το σημείο ενημέρωση όλων των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και ένα ρόλο να διαδραματίσουμε για την ανάπτυξη συνολικής ε, ανάλυσης της έκθεσης ε, ΙΖΑ, τις περίφημες. Είναι ίσως ε, στο άκουσμα λίγο περίπλοκο, αλλά είναι μάλλον απλό. Και με την εμπειρία μου τελευταία 10 χρόνια με καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όταν έχουμε κάποια κρίση, Λαμβάνουμε πληροφορίε από όλε τι πλευρέ. Κάποιε είναι έγκυρε. Κάποιε είναι πληροφορίε οι οποίε στη συνέχεια διαψεύδονται. Σε κάθε περίπτωση όμω υπάρχει τεράστιο όγκο αντικρουόμενων, αντιφατικών συνθήκων. Και η έκθεση λοιπόν αυτή, η ενοποιημένη αυτή έκθεση, είναι απλά μια απόπειρα να οργανωθούν αυτέ οι πληροφορίε και να συλλεχθούν οι πιο ε, επίκαιρε και σωστέ και απαραίτητε πληροφορίε για την ε, κατάσταση. Αυτό ασφαλώ αποτελεί μεγάλη πρόκληση γιατί οι πληροφορίε δεν ε, προέρχονται απαραίτητα από εμά, ε, προέρχονται από πολλά και διαφορετικά σημεία, από τα κράτη-μέλη, από τι οργανώσει, σε διάφορα επίπεδα τη διακυβέρνηση, από τι διεθνεί οργανώσει σε, κάποιες, σε κάποιε περιπτώσει. Και είναι μεγάλη πρόκληση όλα αυτά να συνενωθούν σε ένα κείμενο με τρόπο κατανοητό για όλους. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να ολοκληρώσω στο σημείο εδώ πέρα. Αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για το τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα. Υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου πλέον. Δεν έχει επικληθεί η απόφαση αυτή από κανέναν, αλλά αυτό ασφαλώς μπορεί να αλλάξει ένα πάσα στιγμή. Αν συμβεί κάτι μεγάλο αύριο, μπορεί να γίνει η επίκληση της Ελλήνης Αλληλεγγύης αύριο. Το βασικό μήνυμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα πρέπει να κάνουμε εκπαιδεύσεις, να κάνουμε καταρτήσεις, ασκήσεις, να αναπτύξουμε τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας σε περίπτωση κρίσης και αυτό να γίνεται σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα τα κρατημέλη έχουν εντοπίσει τις σωστές διαδικασίες σε επίπεδο κρατικό για να μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα είναι δυνατή η επίκληση της δεύτερης αλληλεγγύης αν είναι απαραίτητο για να μπορούν να ανταποκριθούν και επαρκώς σε περίπτωση που κάποιος άλλος επικληθεί τη ρήτρα αλληλεγγύη, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τους μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν και μπορείτε σίγουρα να, υπολογίζετε στη βοήθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντάς, λέει η Πρόεδρος. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση δύο γραμματείες θα εξετάσουν ε, το ενδεχόμενο επίσκεψη της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ και του κέντρου ERCC. E Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νίλς Μπράκε. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Αγαπητοί καλεσμένοι. Αρχικά θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή της ε, υπηρεσίας μου, INSEN, γιατί ίσως υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Είναι ο βασικός κόμβος ε, πληροφοριών την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθήκον μας είναι να δίνουμε στρατηγικές αναλύσεις για τους υπεύθυνους χάραξη πολιτική εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε σχέση με την συλλογή προσωπικών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ούτε αξιοποιούμε πληροφορίες για τρίτες χώρες. Οι πελάτες μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και βεβαίως επιμέρους οι πελατε μας ειναι η ευρωπαικη επιτροπη το συμβουλιο τα κρατη μελη και βεβαιως επιμερους οι υπηρεσιες ε, τη ΙΕΣ, του οποίου ήμασταν απόσπαστο τμήμα. Οι εκθέσεις μας βασίζονται σε ε, εθελοντικές ε, συμβολές ε, των κρατών μελών. Δεν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συλλέξουμε μόνιμα στοιχεία πέραν των ανοιχτά διαθέσιμων πληροφοριών που είναι προσβάσιμες από όλους. Ούτε ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τρίτες χώρες. Διαβάζοντα το άρθρο για τη ρήτρα αλληλεγγύης, πρέπει να αναφέρω και ε, Κάποιου περιορισμούς στο ρόλο μας στην εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης. Η ρήτρα αλληλεγγύη στην απόφαση του Συμβουλίου έχει περιοριστεί σε περιστάσεις που ε, λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την επικράτειά της και σε άλλους, ε, άλλες περιοχές δίπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ουσιαστικά Εμάς μας απασχολεί οι ε, στρατηγικές πληροφορίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα τμήμα του οργανισμού μας που αφορά το, την Ευρωπαϊκή Επικράτεια και είναι η, ε, το τμήμα της αντιτρομοκρατίας. Και εκεί έχουμε αξιολόγησης ε, απειλών δεν μπαίνουμε στην ε, αντιτρομοκρατική δράση ούτε με την πρόληψη της τρομοκρατίας ούτε με τα όσα συμβαίνουν εκ των υστέρων μετά από, δηλαδή, από μια τρομοκρατική ενέργεια. Παράγουμε ευρύ φάσμα αξιολογήσεων για τις ε, απειλές και τάσεις της τρομοκρατίας, ιδίως ό,τι αφορά ε, την Ισλαμιστική απειλή στην Ευρώπη, αλλά όχι αποκλειστικά. Η ευρύτερη απειλή καλύπτεται από πολλές θεματικές ε, αναλύσεις στρατηγικών τάσεων και θεμάτων. Όμως εκτάζουμε και ad hoc ε, αξιολογήσεις σε περιπτώσεις ε, τρομοκρατικών ενεργειών. Από εκεί προκύπτει λοιπόν ότι εμείς δραστηριοποιούμεθα με δύο τρόπους. Αφενός συμμετέχουμε την κατάσταση που εγγράφεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4. Μια αξιολόγηση πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου όπως ορίζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη ρήτρα αλληλεγγύη, καταρτίζεται από επιμέρου θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με υφιστάμενου μηχανισμούς. Ένας από αυτού του υφιστάμενου μηχανισμού είναι η ΙΝΤΣΕΝ. Εμεί, λοιπόν μέσω τη ΙΕΣ μπορούμε και συμβάλλουμε σε αυτή την αξιολόγηση της απειλής που δίνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεύτερον, εάν κάποιος επικαλεστεί τη ρήτρα αλληλεγγύης για τρομοκρατική επίθεση στην Ευρώπη, μπορούμε επίσης να συμβάλλουμε στην ε, αύξηση της συνειδητοποίησης και μπορούμε να συμβάλλουμε στην όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων είτε στην Κομισιόν, είτε στο Συμβούλιο, είτε στο κράτος μέλος. Και πάλι σε στρατηγικό επίπεδο. Δεν μπαίνουμε στα ζητήματα της ε, πρακτικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Να κλείσω σύντομα, γιατί καλύτερα να κάνουμε μια συζήτηση Έχω και ορισμένα έγγραφα που μπορεί, μπορώ να σας δώσω αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Ο ρόλος μας έχει περιγραφεί αναλυτικά σε σωρία προφορικών ερωτημάτων του Κοινοβουλίου και έτσι είμαστε διαφανές, ε, διαφανής μηχανισμός. Είμαστε ο μοναδικός υφιστάμενος τέτοιος κόμβος πληροφοριών. Οποιαδήποτε άλλη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών είναι μεταξύ διμερών και πολυμερών συνεργειών. Εμείς ε, δίνουμε ε, τεχνογνωσία και υπερνομοσύνη για πολλές υπηρεσίες που συνεργάζονται στο πλαίσιο της ε, υπηρεσίας μας για να παράσχουμε αξιολογήσεις απειλών υψηλού επίπεδου. Αυτές οι αξιολογήσεις βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη και έτσι Αποκινούμε το στρατητικό σκέλος όπου αυτό είναι απαραίτητο, παράγουμε ολοκληρωμένες τέτοιες αξιολογήσεις ε, απειλών. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήματα. Ευχαριστώ. Να επενθυμίσω ότι ήδη έχει γίνει στο παρελθόν παρουσίαση ε, για το ζήτημα αυτό. Κύριε Μαυρομιχάλη, θα ήθελατε ίσως να παρέμβετε για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Για λόγους πληρότητας και παρότι έχω κάνει την παρουσίαση για τη ρήτρα αλληλεγγύης, θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ στον ρόλο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αλληλεγγύης και ε, η Ίντσεν, όπως είπε ο συνάδελφος Νίλς Μπράκε. Η Ίντσεν λοιπόν είναι αναπόσπαστο τμήμα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Λοιπόν, η ρήτρα αλληλεγγύης, όπως να ακούσατε, είναι τυχόν να αναφερθεί όταν υπάρχει εσωτερική απειλή και καταστροφή στην επικρατειά τους. Όμω η διάκριση μεταξύ εσωτερική και εξωτερική απειλή δεν είναι πάντα τόσο σαφής όσο θα θέλαμε. Γι' αυτό όποτε, όπου δει μάλλον, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος και η υπηρεσία εξωτερική δράσης θα συμβάλλει ακολουθώντας ε, συναφείς ε, πρωτοβουλίες ε, και με βάση τον ε, μέρο διοτήτων της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Όταν υπάρξει επίκληση αυτής της αρχής, θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε τα συναφή και σχετικά μέσα για να επιλύσουμε την κρίση αυτό ενδεχομένω να συμπεριλαμβάνει τον εντοπισμό και προσδιορισμό στρατιωτικών δυνατοτήτων ανταπόκριση σε μια κρίση με τη στήριξη του στρατιωτικού προσωπικού που αποτελεί τμήμα τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση φυσική καταστροφή, οι στρατιωτικέ δυνάμει θα μπορούσαν να συμβάλλουν ε, στην όλη προσπάθεια αντιμετώπιση τη κρίση. Επίσης, έχουμε αυτές τις ε, αναλύσεις ε, Αξιολογήσει απειλών για την διευκόλυνση της λήψη αποφάσεων στο πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όλα αυτά βάσει των πληροφοριών της Ίνσεν και των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά τα συντονίζει το Ευρωπαϊκό Situation Room, που είναι το σημείο επαφή για την υπηρεσία εξωτερική δράση στην περίπτωση ιδιωτική αλληλεγγύη. Εν συντομία, να αναφέρω ότι ότι εκπρόσωπο έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία για να υποβάλει προτάσεις όταν πρόκειται να ζητήσει στρατιωτική παρέμβαση πέραν των ε, συνήθων πρακτικών. Η ρήτρα και ο σχετικός μηχανισμός δεν ε, ενέχει προεκτάσεις για την άμυνα. Δηλαδή, σε περίπτωση που η ανταπόκριση σε μία τέτοια ε, κρίση απαιτεί αντίδραση ECSFP ή CSDP, το Συμβούλιο θα λάβει απόφαση βάσει και των αντίστοιχων ε, διατάξεων ε, της συνθήκης για τις οποίες απαιτείται ομοφωνή γνώμη και απόφαση. Τέλος, να υπογραμμίσω ότι αυτή η απόφαση για τη ρήτρα αλληλεγγύης ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 42.7 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Μαυρομιχάλη. Ο κύριος Μπάρξ έχει το λόγο από το Συνδικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. θα ασχοληθώ λίγο με το μέλλον. Να ρωτήσω κατά πόσον η Εκκλησία Ελληνικής μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση. Το μήνυμά μου θα είναι πως η πολιτική προστασία στην Ευρώπη και ε, ανά την Ευρώπη είναι πάντα ένα θέμα που αφορά τη διεθνή συνεργασία, ειδικά στον ε, περίοδο του ψυχρού πολέμου εξετάζουν την περίπτωση πυρηνικού πολέμου και εξετάζαμε την ε, ανταπόκριση που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε είδους ε, απειλή. Υπάρχουν όμως και Τώρα έχουν προκύψει και η, και η τρομοκρατία. Ε, η ρήτρα λοιπόν αλληλεγγύης θα πρέπει να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Το ερώτημα είναι εάν βρίσκεται στο ύψος των απειλών που δεχόμαστε τώρα και θα ήθελα να εξετάσω συντομία αυτό το ζήτημα. Υποθέτω πως τα τρία πιο σημαντικά στοιχεία είναι ο θεματικός στόχος, ο γεωγραφικός στόχος, σκοπός και ο αυτοματισμός, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει ένας αυτοματισμός στην απάντηση. Το πρώτο θέμα, ο θεματικός σκοπός, θεματικό ζήτημα, τη ρήτρα αλληλεγγύης. Νομίζω ότι το πρώτο θέμα που θα έπρεπε να αναφέρουμε είναι αυτό των σχέσεων με την αμοιβαία υποστήριξη. Το άρθρο 222 αναφέρει ότι η ρήτρα αυτή δεν έχει επιπτώσει στον τομέα της άμυνας, αλλά υπάρχουν δύο άρθρα, το άρθρο 222 και το 427 είναι στενά συνδεδεμένα και το άρθρο 222 αρχικά είχε θεωρηθεί ως μια σύγχρονη απάντηση στις τρομοκρατικές προκλήσεις και απειλές και αφορούσε και την ανθρωπογενή φύση των απειλών τρομοκρατικές οργανώσεις ε, που είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ενώ το 47-2 είναι πιο δύσκολο να ε, ενεργοποιηθεί σε σχέση με το 222 το οποίο δεν είναι και τόσο σαφές. Θεωρώ πως το άρθρο 222 αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις εξάλλου το 122, το 142, το 118 για το ζήτημα του ασύλου και την αλληλεγγύη. Θέματα όπως η μετανάστευση, η ενέργεια γίνονται περισσότερο εδαφικής φύσης πλέον διότι μηχανισμοί όπως αυτός του Δουβλίνου που αφορά στο άσυλο αλλά και στον τομέα της ενέργειας λόγω της ε, κρίσης ε, που σοφεί στις ε, ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τρίτο στοιχείο, το ζήτημα της κλίμακας. Ακούσαμε όλους τους αγορητές που αναφέρθηκαν στο ζήτημα της ε, αλληλεγγύης για να τεθεί σε ενέργεια η ρήτρα αλληλεγγύης πάρθω 41 μάλλον 4-1 το Θεωρώ πως ε, αυτό το οποίο πρόκειται να δούμε είναι συγκεκριμένες απειλές που θα αφορούν στα κράτη. Αυτές είναι τρεις προκλήσεις που βλέπω εγώ σε ό,τι φορά το γεωγραφικό πεδίο. Θα ήθελα να αναφερθώ στην διαχείριση αυτών των απειλών αλλά υπάρχουν διάφορες πτυχές ε, εξοδαφικής φύσης που αφήθηκαν εκτός διαπραγματεύσεων. Το ένα αφορά το ζήτημα των πλοίων υπό ενωσιακή σημαία, το θέμα της πειρατείας, υπάρχει και η εξωτερική κατάσταση, περίπτωση όπου μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα αλληλεγγύης όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δράση μέσω αξιωματικών συνδέσμων και ούτω καθεξής. Ένα τρίτο σημείο αφορά το ζήτημα της εξαγωγής κρίσης. Εδώ, όταν σκεφτούμε την ρήτρα ελεγγύης, έχουμε κατά νου τις καταστροφές που συμβαίνουν στο έδαφος της Ένωσης, αλλά μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση όπου ε, υπάρχει εμπλοκή σε ζήματα μετανάστευσης. Ο ορισμός ε, μιας τρομοκρατικής επίθεσης ε, υπόκειται σε αλλαγές λόγω της ε, χρησιμοποίησης ε, ε, αλλοδαπών και ξένων μαχητών. Υπάρχει επίσης και το ζήτημα της πολιτικοποίησης και μη κρατημέλη τα οποία μετέχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την πολιτική προστασία. Και αυτό λοιπόν μπορεί να ενταχθεί στην τρίτη διάσταση. Και εν συντομία τώρα για το τρίτο επίμεχο ζήτημα που είναι ο αυτοματισμός της ρήτρας αλληλεγγύης ε, Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές πρώτα ανάμεσα στα Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Η Ένωση θέλει να είναι το μυαλό, θα έλεγα, μα, θα έλεγα και αυτή που παρέχει επίσης ε, τα κονδύλια και την ε, νομιμότητα. και μια άλλη διαχωριστική γραμμή Βλέπω ότι ανησυχείτε επειδή έχω μακρηγορήσει. Σταματώ. Σε ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. κύριε Πάξ. Δεν έχουν ζητήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι το λόγο, αλλά παρά όλα αυτά έχουμε κάποιες ε, κάποιους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να ζητήσω από τους πανελίστες μας και ιδιαίτερως ε, όσους εκπροσωπούν τα κράτη, τα, τους δεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας μιλήσουν για την ετοιμότητα το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που γίνει η επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης. Έχουν γίνει ασκήσεις για τέτοια περίπτωση υπάρχει κάποιος ε, μηχανισμός, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την ορολογία γρήγορης αντίδρασης σε τέτοιες περιπτώσεις, στην υποθετική περίπτωση, όπως ε, παρουσίασε η Προεδρία. Πόσο ομαλή θα είναι η χρήση της ρήτρας, λοιπόν. Επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα αυτό. Και τώρα, ίσως κάποιο άλλο ερώτημα. Η κυρία Γκόμες και μετά η κυρία Λούζινγκ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή στον κύριο Ντάς. Πώς εκτιμάει το σχέδιο CRBA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν ε, μάλλον ε, αδύναμη η πρώτη απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ε, εκτίμηση των κινδύνων κτλ. Στη συνέχεια. Κύριε Μπρακ, και εσείς μιλήσατε για το κέντρο ERCC αντιμετώπισης ε, Κρήτης. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει αλληλεπικάλυψη. DG San DG Έχουμε το Sit Vincent. Για βοηθήστε με να καταλάβω. Ποιος ο σκοπός όλων αυτών. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά κέντρα. Μας βοηθάει αυτό τελικά να συντονιστούμε και σε ιδιαίτερα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, γιατί έχουμε δύο κέντρα, το ένα οποίο βασίζεται σε open sources Πείτε μας κι εσείς λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω πώς βοηθάει αυτό. Πείτε μας όμως. Πείτε μας όμως. Εσείς είστε ειδικοί. Εσείς λειτουργείτε τα προγράμματα. στον κύριο Πάρκες ε, ή σε οποιοδήποτε άλλο που θα θέλει να πάρει το λόγο. Αναλύσατε τις συντάσεις που υπάρχουν εντός της ρήτρας αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και επιτροπής. ο ευρυδικός πόλεμος που αντιμετωπίζουμε. Πώς πιστεύετε ότι επηρεάζεται η ρήτρα αλληλεγγύης. Η Ιταλία, για παράδειγμα, τι θα γινόταν αν υπήρχε απειλή από τη Λιβύη, όχι λιβική απειλή, απειλή από τη Λιβύη. Απειλή θα μπορούσε να ζητήσει και να επικληθεί την ε, ρήτρα αλληλεγγύης, για παράδειγμα. Η κυρία Σας ευχαριστώ πολύ. Μία πρώτη ε, ερώτηση προς τον κύριο Πάρξ. Όλο ιδιαίτερος. Μιλήσατε πιο πολύ για τα θεματικά ζητήματα επίκλησης. Και θα ήθελα να στραφώ στην στρατιωτική πτυχή, το στρατιωτικό προσωπικό, τα στρατιωτικά μέσα του άρθρου 222. Στο άρθρο γίνεται ρητά αναφορά ότι τα στρατιωτικά μέσα ανθρωπογενής ε, καταστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μάλλον ε, στρατιωτικά μέσα για ανθρωπογενή καταστροφή. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στα στρατιωτικά μέσα. Από τότε που ε, διάβασα το άρθρο αυτό, Προσπαθώ να καταλάβω τι συμπεριλαμβάνει ο όρος ανθρωπογενείς καταστροφές. Αν αναρωτιέμαι λοιπόν εδώ και χρόνια, κατά πόσον αυτή η ασαφή ε, διατύπωση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε κοινωνικές αναταραχές, για παράδειγμα. Σε μεγάλες, ε, μεγάλα κινήματα διένυξης. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Μίκουτς περιλαμβάνονται και μέτρα ελέγχου εξεγερσεών. Και η προσέγγισή σας για την χρήση αστυνομικών δυνάμεων παρά περίπτωση μεγάλης αντίθεσης και διαδήλωσης του πληθυσμού θεωρείτε ότι είναι σωστή. Οι υπόλοιποι είναι συνάδελφοι από τη Λίμπη. Κορνίλια, έχεις κάποια ερώτηση να θέσεις? Ξέρετε ότι ήταν πάρα πολύ κουραστική ημέρα. Ήταν πραγματικά μεγάλη ημέρα και τώρα α, ακούμε καταστροφές. Α, να ξέρω ότι έχεις και άλλη ερώτηση να κάνεις. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα σώματα, μια από τις πιο μεγάλες επιτροπές νομοφαντικής φύσεως. Η Κορνίλια θέλει να κάνει ερώτηση. Όχι. Κλοντ, τι ερωτήσει που ήθελα να θέσω τις έθεσαν οι συναδελφοί ήδη. Ο κύριο Μπουχνέρ. Ο κύριο Μπουχνέρ Ε, να βγω, δυστυχώ λίγο, αλλά ελπίζω να μην έχουν επαναληφθεί τα ερωτήματα. Μία πρώτη ερώτηση. Αναφέρεται ρητά ότι δεν πρόκειται για αμυντικά ζητήματα, για αμυντικέ υποθέσει. Γιατί λοιπόν το Κοινοβούλιο δεν αναμειγνύεται πλήρω. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε συναπόφαση επί της αρχής, εφόσον πρόκειται για εσωτερικά ζητήματα. Η δεύτερη ερώτηση, όπως ε, ε, η ερώτηση που έθεσε η κυρία Λούζινγκ εδώ στο άρθρο 3α, αναφέρεται σοβαρός αντίκτυπος και μεταξύ άλλων σε ιδιοκτησία. Δηλαδή, μεγάλες κοινωνικές ε, διαδηλώσεις σίγουρα θα έχουν επιπτώσεις σε ιδιοκτησία. Αυτό θεωρώ ότι ανοίγει το δρόμο για καταχρήσεις. Για να μην με παρανοήσετε. Παραβίαση όχι σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, αλλά εδώ πρόκειται για νομοθεσία η οποία υποτίθεται ότι θα είναι στεναρή και θα αντέχει και ενάντια στις αλλαγές και ενάντια στις παραβιάσεις. Επόμενη ερώτηση ότι σε τέτοιες ε, χρήσεις και ασκήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ισχύει το εθνικό δίκαιο, αλλά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η πολύ πιο ασθενής δηλαδή και αδύναμη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ, στο άρθρο 52.3, γίνεται πάλι αφορά στα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και εδώ στο 22 αναφέρεται ότι επιτρέπεται δολοφονία σε περίπτωση ε, που υπάρχει κοινωνική αναταραχή και που είναι απολύτως απαραίτητο. Εδώ και πάλι λοιπόν ανοίγει παρατηράκι για μια μη στρατιωτική επιχείρηση η οποία θα μπορούσε να πάει πάρα πολύ μακριά. Και τέλος, τελευταία ερώτηση. Η ρήτρα αλληλεγγύης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον το ζητήσει η κυβέρνηση του εκάστοτε κράτους. Αλλά στην περίπτωση αυτή τουλάχιστον σύμφωνα με την νομοθεσία, το κείμενο της νομοθεσίας, δεν μπορεί το κράτος μέλος να ε, επηρεάσει πλέον τις δράσεις αυτές. Και ακούσαμε λοιπόν ότι το κέντρο εδώ είναι πολύ ανοιχτό. Μήπως κάνουμε λάθος, αλλά, αλλά από το κείμενο, μόνο βάσει του κειμένου, δεν ε, υπονοείται ότι μπορεί να υπάρχει επιρροή από την ε, κυβέρνηση του εκάστοτε κράτου μέλους που έχει επιτηθεί τη ρήτρα. Μια απάντηση λοιπόν παρακαλώ δώστε μου. Σας ευχαριστώ λέει πρόεδρο να πω ότι κάποια από τα ερωτήματα στράφηκαν σε συγκεκριμένους πανελίστε. Ω εκ τούτου σας ζητώ κύριε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε ξεκινώντας από την Προεδρία. Εντάξει, μπορούμε βεβαίω ε, να ολοκληρώσουμε το δεύτερο γύρο, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Όχι, δεν σα ζητώ δεύτερο ε, γύρο. Απλώ αν είναι ο τελικό γύρο, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ερώτημα. Ξέρω ότι όλοι θέλουμε να πάμε σπίτια μα. Απλώ πολύ σύντομα. Ένα σύντομο ερώτημα για κάποιου συναδέλφου που δεν είναι εδώ Γιατί και άλλοι συναδελφοί ενδιαφέρονται εδώ, και η Κορνίλια, Άννα. Κάτι το οποίο ανακύπτει συνεχώς ε, στο θεματολόγιο της Άμυνα είναι οι αξιολογήσει των απειλών. Θα ήθελα λοιπόν να το θέσω στου συναδέλφου. Κάτι το οποίο θα ήθελα να θέσουν οι συνάδελφοι μου εδώ είναι το εξή. Έχουμε την εντύπωση ότι το Συμβούλιο δεν ξέρει ακριβώ τι κάνει. Να κάνει δηλαδή μία ολοκληρωμένη ετήσια αξιολόγηση και εκτίμηση των απειλών, ούτω ώστε να μα βοηθήσει και όλα αυτά να φτιάξουμε ένα θεματολόγιο άμυνα. Γι' αυτό και εμεί έχουμε ένα ψήφισμα που προτείνει ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον άπαξ ετησίω μια τέτοια εκτίμηση των απειλών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια απάντηση, θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο, γιατί ήταν ένα από τα ερωτήματα που μου έθεσαν κατά τη σύσταση αυτού του ψηφίσματος. Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή αιτήσια αξιολόγηση ή εκτίμηση απειλών. Παρακαλώ, αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα. Να ξεκινήσω με το πρώτο. η αλληλεπίδραση μεταξύ της ρήτρας αλληλεγγύης και του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων του Συμβουλίου. Η διαφορά είναι ότι ο μηχανισμός ηλίτερα αλληλεγγύης έχει εσωτερικό πεδίο εστίασης και μπορεί να επικληθεί κάποιος αυτή τη ρήτρα σε περίπτωση που το κράτος μέλος έχει πληγή σοβαρά και η δυνατότητα ανταπόκρισης δεν είναι επαρκής. Το IVCR, δηλαδή αυτός ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων, αφορά ή μάλλον παρέχει μία πλατφόρμα ειδικά προσαρμοσμένης και ταχύτητας ανταπόκρισης σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την κρίση, είτε αυτή η κρίση είναι εντός είτε εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Έτσι αυτός ο μηχανισμός μας βοηθά να δομήσουμε κάπως αυτή την ανταπόκριση. Και όταν γίνεται επίκληση της αρχής της ελεγγύης. Δηλαδή αυτός ο μηχανισμός του, του Συμβουλίου αυτομάτως τίθεται σε λειτουργία από την Προεδρία. Για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όταν εξετάσαμε τη μορφή που θα πρέπει να πάρει η απόφαση του Συμβουλίου, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης και ποιες είναι οι καλύτερες διαδικασίες. Προσπαθήσαμε βεβαίως να επιτύχουμε συμβασμό μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και ΕΕ η εκπροσώπου. Κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποκλείεται το Κοινοβούλιο σε καμία περίπτωση. Η Προεδρία ενημερώνει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό δεν είναι μόνο από ευγένεια. Και εγώ θέλω να τονίσω ότι πρέπει να εργαζόμαστε από κοινού σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Επομένως, όπως έχει κάνει και το Κοινοβούλιο σε άλλες κρίσεις, μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε σε ό,τι αφορά την διαφάνεια, την προβολή, το πολιτικό σας βάρος, ακόμα και με οικονομικούς πόρους ενδεχομένως, για να μετριαστούν οι επιπτώσεις ε, των κρίσεων. Επομένω, και εμείς ε, βασιζόμαστε και στη δική σας ε, συνδρομή και αρρωγή. Ενδιαφέρον ερώτημα ακούσαμε και για τον υβριδικό πόλεμο και τη δυνατότητα επίκλησης της ε, ρήτρες αλληλεγγύης ή αμοιβαία άμυνα. Ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αλληλεγγύης, κατά τη γνώμη μου, ή τουλάχιστον το πώς έχει διατυπωθεί στην ε, συνθήκη. Από την πλευρά της πρόληψης, αυτό ισχύει μόνο για, την, ε, για τις τρομοκρατικές απειλές και άλλες, ή άλλες ή μάλλον φυσικές καταστροφές. πρόκειται μόνο για ανταπόκριση. Για τις υβριδικές απειλές, ίσως βεβαίως να πρέπει να υπάρξει σε βάθος ανάλυση αν το χρόνο, όμως είναι ενδιαφέρον το ζήτημα. Για τις αξιολογήσεις των απειλών που αναφέρατε, μπορώ σχεδόν να παραθέσω ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι αυτό εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εάν δηλαδή οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων αποφασίσουν ότι απαιτείται ανάλυση και εκτίμηση ενός συγκεκριμένου κινδύνου μιας απειλής, τότε δίνουν αυτή την εντολή και όλα τα διαφορεμένα μέρη βεβαίως συνέρχονται και παίρνουν τις απαραίτητες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντάς. Ευχαριστώ. Ορισμένες παρατηρήσεις από πλευρά μου. Αρχικά προς το ερώτημά σας, κατά πόσο είμαστε έτοιμοι, αν είναι σε ετοιμότητα οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Πολλά έχουν γίνει, πιστεύω, και ήδη έχουμε αποκομίσει πείρα μέσω των διαφόρων μηχανισμών και εργαλείων από πλευρά πολιτική προστασία. Κάνουμε πολλά σεμινάρια κατάρτιση, δοκιμές, ασκήσει με τα κράτη-μέλη. Πρόσφατα είχαμε και, μία, και ένα πρόγραμμα προετοιμασία σε διάφορα στάδια που είχε προετοιμάσει η Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων. Και το πρόγραμμα ΡΕΤ που ήταν ε, ε, πλήρους κλίμακας ε, σε περιπτώσεις ομοιρίας σε περιβάλλον CBRN. Έχουν λοιπόν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση της ετοιμότητας. Για να δούμε και πώς εντάσσεται και η ρήτρα της αλληλεγγύης όλα αυτά. Όμως συμφωνώ ότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν και αυτό είναι κοινή πρόκληση για όλους και πρέπει στα επόμενα χρόνια πραγματικά να επενδύσουμε σε αυτόν τον τομέα, να αυξήσουμε την ετοιμότητα και να λειτουργήσει στην πράξη αυτή η ρήτρα αλληλεγγύης. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν ε, αυτοσχεδίως κατά τη διάρκεια μιας ε, κρίσης. Πρέπει να τα έχουμε προβλέψει από πριν. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν με βάση πρώτερου σχεδιασμού και όχι εκείνη τη στιγμή αυθορμήτως. Πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων τι θα κάνει ο καθένας, τι θέτουμε ως προτεραιότητες και το καθεξής. Ο σχεδιασμός λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικός. Πρόσφατα, να, συγγνώμη, σύντομα να απαντήσω στην κυρία Γκόμες. Δεν ε, πρόκειται να κάνω κάποια εκτίμηση του προγράμματος CBRN, όμως συμφωνώ ότι πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν για την αύξηση της τιμότητάς μας σε τέτοιου είδους ε, κινδύνων, πυρηνικών, βιολογικών όπλων, πυρηνικών όπλων. Αναπτύσσουμε ένα μηχανισμό ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει τη μορφή ενός ε, ε, εθελοντικού μηχανισμού που θα μπορούν να αναπτύσσουν τα κράτη-μέλη, τις δυνατότητές τους για κοινέ επιχειρήσεις σε περιπτώσεις κρίσεων και νομίζω ότι το CBR είναι ένας τομέας που θα πρέπει να αναπτύξουμε σε αυτό το πλαίσιο. Στο σημερινό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο ε, είναι ανούσιο όλα τα κρατημέλη να επενδύουν σε ακριβώς τις ίδιες ε, ενέργειες και τεχνολογίες. Πρέπει από κοινού να εργαστούμε και να αναπτύξουμε συγκεκριμένες μορφές ανταπόκρισης σε περίπτωση κρίσεων, βάσει κατάλληλης αξιολόγησης απειλών και να υπάρξει συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Επομένω, μπορούμε να κάνουμε πολλά για να προετοιμαστούμε και τέτοιου είδου απειλέ. Έχουμε επίση τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μία δυνατότητα, ένα μηχανισμό ανάσχεση, buffer capacity, κάτι το οποίο δεν ε, χρειαζόμαστε πολύ συχνά, αλλά και πάλι πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει οικονομική αιτιολόγηση οποιαδήποτε για να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους μηχανισμούς και στα 28 κράτη-μέλη. είναι θέμα κοινή λογικής και οικονομικού συμφέροντος να επενδύσουμε από κοινού τέτοιου πόρου για τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίε. Και τέλος, για τον πολλαπλασιασμό των κέντρων και πάλι ε, θίγεται κάτι το οποίο είναι σημαντικό θέμα, όμως θέλω να το θέσω στην κατάλληλη διάσταση. Ε, στην Επιτροπή σήμερα έχουμε τρία ουσιαστικά ε, κέντρα κρίσεων. ERCC, το κέντρο συντονισμού δηλαδή ε, κρίσεων στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, ε, κέντρο κρίσεων στη DG Home, που αφορά κυρίως τα ζητήματα της ε, Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων, που αφορά κυρίως την προστασία, δηλαδή είναι διαφορετικό από το ERCC. Μετά στη ΣΑΝΤΕ έχουμε μηχανισμό κρίσεων σε ό,τι αφορά την, ε, η δημόσια υγεία πιο συγκεκριμένα. Δεν διαφέρει πολύ από τα όσα βλέπετε και στα κρατη Και στα κρατη δηλαδή, οι επιμέρους αρχές θα έχουν το δικό τους κέντρο από το οποίο συντονίζουν ε, την ανταπόκρισή τους. Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν δικό τους κέντρο, η πυροσβεστική έχει διαφορετικό κέντρο, ε, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει άλλο κέντρο, αυτή η συνύπαρξη λοιπόν δεν δημιουργεί απαραίτητα κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει μάλιστα ένα πλεονέκτημα ε, του να έχουμε την αντιμετώπιση της κρίσης κοντά στον τομέα πολιτικής που μας αφορά και έτσι οι ειδικοί αναλαμβάνουν την κρίση. Και έτσι υπάρχει στενή ε, διασύνδεση μεταξύ αντιμετώπισης κρίσης και του τομέα πολιτικής. Τούτου λεχθέντος νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει πολύ σημαντική προσπάθεια ε, ανάπτυξη της μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ επιμέρους ε, κλάδων. Θέλουμε να αναπτύξουμε το ε, κέντρο συντονισμού ανταπόκρισης κρίσεων ως ε, κύριο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων. Το ERCC λοιπόν έχει συνάψει μνημόνιο κατανόηση με όλε τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω κάτω και έτσι προσφέρουμε κάποιε οριζόντιε υπηρεσίε σε όλε τι υπόλοιπε υπηρεσίε ό,τι αφορά τι πληροφορίε, δορυφορικέ εικόνε, συντονισμό και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε κάποιε τέτοιε λειτουργίε που άφτονται τη αντιμετώπιση κρίσεων στο ERCC. Έχουμε και δικό μα σύστημα μέσα από το οποίο συντονίζουμε ε, τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από όλες τις επιμέρους ε, υπηρεσίες της Κομισιόν κατά τη διάρκεια κρίσεων και εκεί το ERCC θα είναι βασική πλατφόρμα που θα στηρίζει ε, το συντονισμό. Νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για τον εξορθολογισμό αυτού του ζητήματος και νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι στην οργάνωσή μας. Ευχαριστώ κύριο Σμπράκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να διευκρινίσω το εξής. Το Ίνσεν είναι το καινούργιο όνομα του Ζίτσεν. Το παλιό Ζίτσεν αποτελούταν από το τμήμα της ανάλυσης και ε, το Situation Room. Έχουμε λοιπόν τώρα το Ίνσεν, το οποίο αποτελεί βασικά το τμήμα της ανάλυσης και έχουμε και το Duty Area, το Situation Room, το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος, το οποίο βρίσκεται σε διαφορετικό τμήμα του κτηρίου. Εμείς κάνουμε την ανάλυση ενώ το Situation Room ουσιαστικά καταγράφει τα γεγονότα. Σε ό,τι αφορά το Open Sources, είναι ένα κοινό μυστικό ότι σήμερα το έτος 2015 μία σειρά εκθέσεων μυστικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν επίσης open source. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος της συλλογής πληροφορίας. Οι μυστικές ε, πληροφορίες και υπηρεσίες δραστηριοποιούνται μετά. Ακούμε τις ειδήσει, βλέπουμε τι γίνεται και μετά μόνο μπορούμε να πούμε στις μυστικές υπηρεσίες να κάνουν ανάλυση. Άρα ναι, το open source ε, το έτος 2015 αποτελεί σημαντικό στοιχείο οποιαδήποτε τέτοια ανάλυσης. Άκουσα μια δεύτερη ερώτηση για τον υβριδικό πόλεμο. Θα μπορούσα λοιπόν να φανταστώ μια μεγάλη επίθεση στα συστήματα IT, ξέροντας πόσο εξαρτώμαστε από τα συστήματα IT πλέον και είναι και θέμα φυσικά ορισμού, αλλά αν ένα μεγάλο σύστημα IT σε ένα κρατός μέλος ε, έμπαινε στο στόχαστρο της επίθεσης, θα μπορούσε να επικληθεί ρήτρα ελεγγύης. Για το στρατιωτικό, την χρήση στρατιωτικών δυνάμεων και για την ε, αρμοδιότητα ε, της Εθνικής Αρχής και του Εθνικού Δικαίου. Δεν υπερσκελίζεται το Εθνικό Δίκαιο. Το κράτος μέλος επιλέγει να επικληθεί τη ρήτρα Δεν μπορεί να επιβλεφθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος α, Τα άλλα κράτη δε δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα στο κράτος χωρίς την θέλησή του. Και οποιαδήποτε δράση στο κράτος μέλος θα πρέπει να βασίζεται στην νομοθεσία του εκάστοτε κράτος μέλος. Δεν ε, είμαστε, είπα, που υπάρχει ομοσπονδιακό νομοϊκό σύστημα. Δεν υπάρχει ομοσπονδιακό σύστημα. Δεν υπάρχει ομοσπονδιακή αστυνομία. Ούτε FBI μπορούμε να φτιάξουμε. Δεν υπάρχει ομοσπονδιακή εισαγγελία, ομοσπονδιακό ποινικό δίκαιο, ομοσπονδιακή δίωξη. Δεν υπάρχει ομοσπονδιακό στρατιό. Αν αποστείλουμε μαχητέ ή, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε υπηρεσία κατεπίγουσα ανάγκη, στην Πεσίβιου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την Ιταλία για το Βεζούβιο, το παράδειγμά σας, θα πρέπει να βρουν σύμφωνα με το Ιταλικό δίκαιο και υπό την Ιταλική κυβέρνηση. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω γιατί στο παράδειγμά σας οι 150 νόμοι που χρειάστηκε να αλλάξουν. Ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον χρειάζεται πιο πολλές ε, διμερείς ε, συμφωνίες για να μπορούν τα εργαλεία και οι υπηρεσίες προστασίας των πολιτών να μπορούν να δρουν στις χώρες. Ένα παράδειγμα, αν υπάρχει η χρήση αστυνομικών δυνάμεων για το ποτόσφαιρο. οι αστυνομικοί πηγαίνουν ε, μαζί με τους οπαδούς από το ένα κράτος στο άλλο. Για να γίνει αυτό όμως που γίνεται, ε, υπάρχουν εκτενείς διμερείς ε, συμφωνίες. Γιατί για να υπάρξει και να έρθει η αστυνομία στην Ολλανδία, για παράδειγμα, σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, θα πρέπει αστυνομικό, από που και αν είναι, να τηρεί το Ολλανδικό δικαίωμα. Το στρατιωτικό προσωπικό, τι μπορεί να κάνει το στρατιωτικό προσωπικό. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαμε υπόψη μας κατά την ε, κατάρτιση του κειμένου το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά μιλάμε για εργαλεία, για βιολογικές, χημικές επιθέσεις και συχνά α, τα εργαλεία αυτά, τον εξοπλισμό αυτών, τον έχει στα χέρια του ο στρατός. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτόμαστε και αναφέρεται το στρατιωτικές δυνάμεις για τις ε, ετήσιες αξιολογήσεις και εκθέσεις ε, κινδύνου. Να σας πω ότι υπάρχουν ήδη τέτοιες εκθέσεις. Ε, η έκθεση οργανωμένου εγκλήματος, η, έκθεση για, το για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εμείς ε, είμαστε έτοιμοι να καταρτήσουμε οποιαδήποτε έκθεση μας ζητηθεί ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, και τώρα το λόγο έχει ο κ. Πάρξ. Καταρχήν μας κ. Λούζινγκ, οι εφαρμοστικές αποφάσεις ε, μιλάνε πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί τα εθνικά μέσα που είναι διαθέσιμα. Τώρα, η υπέρβαση ζήλου, ο υπερβολικός ζήλος μάλλον, δεν θα πρέπει να προκαλεί κάποιες ε, κοινωνικές εντάσεις ε, όπως ε, το παράδειγμα της Πορτογαλίας της Ελλάδας κάποιο κράτος μέλος χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια Τώρα για τους στρατιωτικούς πόρους η διάκριση ανάμεσα σε πολιτικές και στρατιωτικές, ε, πολιτικούς και στρατιωτικούς ε, πόρους ε, δεν είναι πάντα εύκολα διακριτή. Δεν θέλαμε να γίνει μια επαναστατικοποίηση, θα έλεγα, των μέσων. Να υπάρχει το θέμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αστυνομίας Χορφυλακής τώρα για τον Ιδρυτικό Πόλεμο Λιβύη κλπ. Πρέπει να αναρτηθούμε πόσες ε, πιθανότητες υπάρχουν για έναν παρομοιβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη. Όταν ένα κράτος μέλος το θίξει, θα χρειαστεί να γίνει μια πολιτική ανάλυση πάνω στο ζήτημα. Κατά πόσο δηλαδή μια ρήτρα αλληλεγγύης μπορεί να αποτελέσει στο κάτω κάτω και μια πρόκληση. Δεν έχω απάντηση, δεν έχω και μια παρόμοια ανάλυση. Αλλά υπάρχει δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, πολλά ζητήματα που άπτονται της ρήτρας ε, αλληλεγγύης και της ρήτρας αμοιβαίας ε, αρρωγής ε, είναι ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή η ακρόαση δεν αποτελεί μια ακαδημαϊκή νομική συζήτηση, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πολιτικό στοιχείο Κύριε Συμπρόεδρε, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω γιατί πιστεύω, όπως είπαμε σήμερα το πρωί, σε μια κοινή αχρόαση με την ίντα, είναι πραγματικά ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας, παρά το γεγονός ότι μόνο δύο θαραλέοι συνάδελφοι έχουν μείνει μέχρι τελική πτώσεως. Ο, ο, πάντα, πάντα είναι ένας αγώνας κατά του χρόνου γιατί σωματικά δεν είναι δυνατόν να είμαστε παντού και καταλαβαίνουμε ότι οι συνάδελφοι έχουν υποχρεώσει. αλλά νομίζω ότι στην αρχή πολλοί συνάδελφοι από τη ΛΥΜΠΕ ήταν εδώ. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι διοργανώνονται αυτές. Καταλαβαίνετε βέβαια, καταλαβαίνετε και το εκτιμάμε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μας ενδιαφέρει και θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή. Την εκτιμούμε ιδιαίτερως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέκη Πρόεδρος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η δημόσια ακρόαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους μας τους πανελίστες για τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω και στα μέλη της Επιτροπής ΕΝΤΕ. Αύριο ξεκινάμε στις 10.30. και θα τελειώσουμε την ίδια ώρα. Α, το απόγευμα θα είναι ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση. Θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο μαζί με δύο άλλες επιτροπές από κοινού. Ευχαριστώ πολύ.